So good afternoon everyone. First of all... Γεια Καλησπέρα σε όλους σας. Πρώτο, ανακοινώσεις. Έχω την εξή ανακοίνωση να σας κάνω. Έχουμε λετονική διερμηνία για τη συζήτηση αυτή. Προφανώς έχουμε ε, διερμηνία στα λετονικά και ευχαριστώ τις υπηρεσίες διερμηνίας που απέντησαν τόσο γρήγορα και τόσο εύστοχα. Και περνούμε μέσω στο σημείο 9 λοιπόν, η εθέτηση του ευρώ από τη Λετωνία την 1η Ιανουαρίου του 2014 είναι η έκθεση Μπάλτς. Δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι από πλευράς μου διαπίστωσα ότι έχει κάνει αξιοθαύμαστη πρόοδο η Λετωνία τα τελευταία χρόνια. Το 2008 ξέρουμε ότι την έπληξε ραγδαία η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και αποτέλεσμα ήταν η οικονομία της να, να βυθιστεί σε πάρα πολύ βαθιά κρίση. Δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα ε, ως γνωστό δόθηκαν δισεκατομμύρια συνολικά τα κονδύλια 4,5 δις. Μέσα σε τέσσερα χρόνια η λετονική οικονομία ανέκαμψε θαυμάσια και σήμερα είναι και υποδειγματική χώρα και παράδειγμα που χρησιμοποιεί κανείς για το πώς η λιτότητα και τα μέτρα εξοικονόμησης μπορούν να υπερβούν την κρίση. το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που πληρώθηκε στο δάνειό του και νωρίτερα μάλιστα και επίσης ε, τα χρήματα που οφείλονται στην Παγκόσμια Τράπεζα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση του χρόνου θα έχουν αποσβεστεί. Η χώρα λοιπόν έχει αυτή τη χαρμόσυνη εξέλιξη πίσω της και από ό,τι μου φαίνεται εμένα ως εισηγητού είναι λογικό να μπει στο ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνει πολλή δουλειά ο λαός της Λετωνίας. Τέλη Μαΐου Είχα την ευκαιρία να αποκομίσω ιδία άποψη, πήγα για ένα τριήμερο ε, μετά από ε, πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας επισκέφθηκα την πρωτεύουσα τη Ρήγα. Μου έκανε εντύπωση η βούληση και οι προσπάθειες των αρμοδίων αρχών και της κυβέρνησης για να ετοιμαστούν για το ευρώ. Κατά τη διάρκεια της επισκεψής μου, θέλω να το πω και αυτό ξεκάθαρα, δεν μίλησα μόνο με εκπροσώπους της κυβέρνησης, ε, της οικονομίας, των τραπεζών και των ασφαλίσεων, αλλά ακριβώς, γιατί είχα ιδιαίτερη επιθυμία γι' αυτό, ήρθα σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών αλλά και οργανώσεις που σαφώς είναι κατά της ένταξης ε, στο ευρώ της Λετωνίας. Και αυτές ακριβώς οι συζητήσεις ήταν άκρως ενδιαφέρουσες και μου έδωσαν και μια νέα εικόνα και την ατμόσφαιρα γενικά γύρω από την εισαγωγή του ευρώ στη Λετωνία. Και το εξής έγινε αμέσως σαφές και πολύ γρήγορα. Οι περισσότεροι Λετωνοί απομένουν ακόμα να πιστούν για την είσοδο στο ευρώ. Η κυβέρνηση της Λετωνίας θα πρέπει να δουλέψει σκληρά για την επικοινωνία και την ε, ενημέρωση, γιατί για μένα η μεγαλύτερη ανησυχία μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα επαρκής αποδοχή από τον πληθυσμό για να το διατυπώσω έτσι προσεκτικά. Στις συζητήσεις που είχα επιτόπου φάνει ξεκάθαρα ότι πολλοί είναι εκείνοι οι πολίτες στη χώρα που δεν αισθάνονται παρκώς ενημερωμένοι για να κάνουν έναν επικοδομητικό και εκτενή διάλογο με τις αρχές, των οποίων και επιθυμούν όμως. Μετά παίζει μεγάλο ρόλο ο κίνδυνος ότι θα χάσουν την ταυτότητά τους και ότι θα πάνε στα ύψη τιμές. Και σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ε, έτσι, η αρνητική ατμόσφαιρα διορθώνεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού είναι υπέρ της εισαγωγής του ευρώ μέχρι τώρα και κατά την άποψή μου, όπως σας είπα, παραμένει χαμηλό αυτό το ποσοστό. Ε, τώρα, ε, οι επίσημες εκστρατείες ενημέρωσης και πληροφόρησης είτε ήδη έχουν ξεκινήσει, ε, είτε θα αρχίσουν και μετά την τυπική και επίσημη απόφαση όταν ληφθεί αυτή. Και εδώ νομίζω ότι χρειάζονται κάποιες προσαρμογές. Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος τώρα θα πρέπει να φτάσουμε σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στην Ήπεθρο και να ενημερωθούν για το ευρώ εκτενώς και συνολικά και με τρόπο εύληπτο και κατανοητό. Εγώ είμαι αισιόδοξο, αγαπητοί συνάδελφοι. Με ένα ναι των Βρυξελών μπορεί να σταλεί ένα θετικό μήνυμα και να αυξηθεί και η αποδοχή στον πληθυσμό και τους επόμενους μήνες μέχρι την ημερομηνία ένταξη στο ευρώ. Τώρα, τα κριτήρια σύγκλησης, επιτρέψτε μου δύο λόγια για αυτά. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι πληρούνται τα κριτήρια. Άλλωστε αυτό το μαρτυρούν και εκθέσεις Κεντρικής Τράπεζας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση μόνο. Τα σημερινά αριθμητικά στοιχεία της ΕΚΤ και της Κομισιόν είναι εύγλωτα και δείχνουν μια εικόνα αρκετά αισιόδοξη για την κατάσταση της λετωνικής οικονομίας και ως προς τη βιωσιμότητα της σύγκλησης. <laughs> για τη σταθερότητα των τιμών, ο πληθωρισμός είναι 1,3% και είναι κάτω από τα τρία κράτη αναφοράς που είναι 2,7 γνωρίζουμε ο πληθωρισμός τώρα και οι άλλες δύο χώρες είναι η Ιρλανδία και η Σουηδία. Τα δημόσια οικονομικά βεβαίως είναι θετικά. 1,2% είναι μόνο το έλλειμμα του προπολογισμού, το χρέος 40,7% τέλη του 2012 και αυτό είναι ένα κριτήριο πάρα πολύ ευπρεπές τα μακροπρόθεσμα επιτόκια 3,8% και εδώ πάλι είναι κάτω από τα τρία ε, κράτη αναφοράς. Είναι πάρα πολύ θετικά όλα αυτά τα στοιχεία για την οικονομία, τα αριθμητικά. Επιτρέψτε μου τώρα μερικά ακόμα σχόλια. Ακούστηκαν επιφυλάξεις στο παρελθόν για τη στιβαρότητα του τραπεζικού τομέα είναι περίπου 50% οι ξένες καταθέσεις εκεί σε σχέση με το σύνολο. Ε, ο τραπεζικός τομέας στη Λετωνία σίγουρα με ευρωπαϊκούς όρους είναι μικρός, 130% του ΑΕΠ σε σύγκριση με την Ένωση που είναι 370% ε, περίπου. Ε, οπότε αυτό το φαινόμενο με τις ξένες καταθέσεις δεν είναι καινοφανές, το αντίθετο. Ε, είναι μακρά η παράδοση στη Λετωνία ε, ότι κάνει ε, business με ξένες καταθέσεις και αυτό εξηγείται και πολιτιστικά και ιστορικά και γεωγραφικά. Γιατί υπάρχει μεγάλη ρωσόφωνη μειονότητα στη χώρα. Οι τράπεζες που κατά κύριο λόγο έχουν ξένες καταθέσεις, έχουν αυστηρό έλεγχο πολύ πιο αυστηρό από άλλες τράπεζες, ακριβώς ε, για να αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι. Αυτό συζητήθηκε ε, και με την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς της Λετωνίας, που είναι αρμόδια για την τραπεζική εποπτεία και επίσης με εκπροσώπους των ιδίων των τραπεζών. Οπότε μπορώ να σας πω και να σας βεβαιώσω ότι υπάρχει πολύ ενεργή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των ελόγων τραπεζών ακριβώς για να περιορίζονται και να αποφεύγονται και να αποσοβούνται οι κίνδυνοι. Βεβαίως δεν θέλω να υποτιμήσω τον εδεχόμενο κίνδυνο, το πιθανό αυτών των ε, τραπεζών. Ε, θα πρέπει να συνεχιστεί ε, ενεργά και ο έλεγχος και η παρακολούθηση και η υποπτία των τραπεζών αυτών. Κατά την άποψή μου η Λετωνία δεν μπορεί να συγκριθεί με την Κύπρο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι συγκρίση με την Κύπρο. Είναι τελείως διαφορετικές οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες. Γιατί έχω ακούσει σε μεμονωμένες συζητήσεις διάφορα. Κατά την άποψή μου δεν συγκρίνονται, είναι ανώμια τελείως τα συστήματα. Τέλος. Για ποιο πράγμα ανησυχώ η ενέργεια παραμένει ψηλή. Τέλη του 2012 ήταν 15% και ιδιαίτερα οι περιφερειακές διαφορές και ε, μη προσαρμογή ορισμένων τομέων είναι προβληματική και έχουν να κάνουν και καθορίζουν το μεγάλο σχετικά αριθμό του επίπεδου της ενεργείας. Γι' αυτό θα πρέπει οι διαρθρωτικές ελλείψεις στην αγορά εργασίας θα πρέπει να ξεπεραστούν με μια πιο ενεργή πολιτική, πιο δραστήρια και μια μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού κατά την άποψή μου συστήματος. Συνοψίζω. Η εκτίμηση μου είναι ω εξής. Έχει περάσει πολύ σκληρή ρητότητα και σκληρές μεταρρυθμίσεις η Λετωνία για να βγει από την κρίση και το λέω και ως εισηγητής του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής και μια αναγνώριση, αλλά υπήρχε και κόστος ε, που είναι οι μεγάλοι δείκτες ανεργίας που παραμένουν, ε, οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθούν για να είναι βιώσιμη η εξέλιξη της ε, οικονομίας και να είναι βεβαιωμένη και η τήρηση των κριτηρίων σύγκλησης. Τελευταία πρόταση Πιστεύω ότι η Λετωνία βρίσκεται στο σωστό δρόμο και το ευρώ θα βοηθήσει ε, τη χώρα να σταθεροποιηθεί έτσι περαιτέρω και καλωσορίζω ρητά και θερμά την εισδοχή της χώρας στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. John, the Τώρα θα δώσω το λόγο στους σοσιαλιστές και θα τους εκπροσωπήσει ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκπροσωπώ το σκιώδη μας συγητή, δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Θα σας παρουσιάσω την αποψή του λοιπόν. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αντικειμενική και ισορροπημένη έκθεση. Σημείωσε τις προσπάθειες που έκανε ο λετωνικός λαός και η λετωνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια που ήταν αξιοσημείωτες. Όχι μόνο ισοσκέλισαν τους λογαριασμούς τους, αλλά ξανά βάλαν την οικονομία σε θετική τροχιά. Είναι από τους πρωτοπόρους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Αλλά κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις και μην ξεχνάμε λοιπόν και τους πιθανούς κινδύνους. Να αναφέρω μερικούς που καλύπτει και η έκθεση ούτως ή άλλως. Καταρχάς η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και το μερίδιο που έχουν οι καταθέσεις των μη κατοίκων, των μη μεδαπών. Ε, λόγω πολιτιστικών και γεωγραφικών λόγων ε, ελήφθησαν μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος ε, λόγω αυτής της κατάστασης. Υπάρχει ο πολιτικός κίνδυνος, είναι πολύ σημαντικό για τη Λετωνία και το μέλλον της Ευρωζώνης η χώρα να παραμείνει σε μια συνετή πολιτική τροχιά και να μην προσπαθήσει να βρει έτσι βραχυπρόθεσμες μαγικές λύσεις. Θα πρέπει να υπάρξει διαφανεία Αναφέρομαι στην τιμή του ρυζιού εδώ που έχει αυξηθεί υπερβολικά. Είναι πολύ σημαντικό, να, όπως είπε και ο εισηγητής, να έχουμε σωστές εκστρατείες πληροφόρησης. Επίσης, η διαρθρωτική ανεργία. Ε, ο εισηγητής μιλάει για μεταρρύθμιση της εκπαίδευση και της αγοράς εργασίας. Με βάση τα θετικά που παρουσιάζουν όλοι οι τομείς, ο κ. Παγκάρ εκ μέρους των σοσιαλιστών υποστηρίζει και την έκθεση και την ένταξη της Λετωνίας στην Ευρωζώνη. Εγώ προσωπικά θέλω να επιβεβαιώνω αυτά που, επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο σκιώδης συγητής μας, να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις της Λετωνίας και τέλος να καλωσορίσω την Λετωνία ε, στην Ευρωζώνη. Σας ευχαριστούμε κύριε Κούτας. Και τώρα ο κύριος Κλίντ από τους φιλελεύθερους. Ο κύριος Κλίντ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, καταρχάς, οι δύο προλαλήσαντες ανέφεραν τα σημαντικά σημεία. Λίγα έχω να προσθέσω εγώ μόνο. Όλοι γνωρίζουμε ότι ακριβώς η σχέση του πληθυσμού, του λαού με το νόμισμα είναι καθαρά ψυχολογική σε μεγάλο βαθμό. Οπότε δεν θα πρέπει να το υποτιμούμε ότι δύο τρίτα ακόμα των λετωνών είναι πολύ προσιλωμένοι στο νομισμά τους και έχουν πολύ επικριτική στάση απέναντι στο ευρώ. Και θα είναι πάρα πολύ αποφασιστικό το εξής. Το πρώτο χρόνο ή την πρώτη διετία θα πρέπει να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης στο λαό. Δηλαδή με την έλευση του ευρώ θα παραμείνει το νόμισμά τους σταθερό και δεν θα οδηγήσει σε ε, πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές. Γνωρίζουμε από ίδια πείρα από διάφορα κράτη ότι παντού έταξαν όλοι τα ίδια, αλλά τηρήθηκαν σε ελάχιστε περιπτώσεις αυτές οι υποσχέσει. Μπορώ να σας πω στη δική μου χώρα τι έγινε. Τα ίδια μας έλεγαν, αλλά de facto οι τιμέ πήγαν στα ύψη και μάλιστα και στις υπηρεσίες πάρα πολύ ψηλά και πολύ γρήγορα. Αυτό θα πρέπει να αποφευθεί οπωσδήποτε, αλλιώς θα απογοητευτεί ο λαός. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και τους πιθανούς κινδύνους και να τους έχουμε υπόψη μας. Για τις ξένες καταθέσεις έγινε λόγος, δεν έχω να προσθέσω τίποτα, αλλά εγώ θεωρώ έναν άλλο παράγοντα επικίνδυνο. Είδαμε τι έγινε με τη Λιθουανία που το 2006 του 2007 παρά λίγο να μπουν στο ευρώ τελικά δεν το έκαναν γιατί υπήρχε αβεβαιότητα ως προς τον πληθωρισμό. Εδώ νομίζω είναι αντίστοιχο το θέμα της ενέργειας. Η Λετωνία εξαρτάται από εισαγωγές ενέργειας και ε, πάρα πολύ ακόμα από τη Ρωσία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και οι εξελίξεις ακριβώς αυτό το τομέα και των τιμών μπορεί να ε, ενέχουν διάφορους κινδύνους, υποθέσεις και ε, τα διάφορα δεδομένα που έχουμε στο μυαλό μας να ανατραπούν. Και θα πρέπει λοιπόν και ποσοτικά να έχουμε... Ποιο θα ήταν το ε, ρίσκο, ας πούμε. Αν αυξηθεί κατά 20% η τιμή της ενέργειας, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό και στην εθνική οικονομία αλλά και στο λαό γενικά. Ε, ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι για μας, για τα 17 κράτη του ευρώ, της Ευρωζώνης, είναι μεγαλύτερη επιτυχία να μπει η, Ευρω... Λετωνία στο ευρώ παρά για την ίδια τη Λετωνία. Γιατί αυτό δείχνει ότι ε, παρόλε τι δυσκολίε υπάρχουν λαοί και χώρες που πιστεύουν στο ευρώ και θέλουν να ενταχθούν και ενδιαφέρονται. Βέβαια, δεν θέλω να σα κρύψω ότι για τους Λετωνούς είναι πάρα πολύ πολιτική απόφαση, διότι αν μπουν στη λέσχη του ευρώ, στην ευρωζώνη, τότε συνδέονται ακόμα περισσότερο με τις χώρες κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης από ό,τι είναι μέχρι τώρα και αυτό είναι και συμφέρον τους γενικά. Συμπέρασμα, ε, θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε με αυτά που είπαμε. Ευχαριστώ κύριε Κλίντς ε, από τους Πρασίνους. Το λόγο έχει ο σχεδοσηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εμείς ε, διατρανώνουμε την υποστήριξή μας. Είμαστε πολύ θετικοί στην είσοδο της Λετωνίας στην Ευρωζώνη στο βαθμό που είναι ένα επιπλέον μήνυμα αυτό, ένα επιπλέον σημάδι ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και το έχουμε ανάγκη αυτό σε αυτή την ε, περίοδο που βιώνουμε. Γι' αυτό ακριβώς υποστηρίζουμε το ψήφισμα που μας προτείνει ο συγητής μας, ο οποίος εξάλλου έχει δίκιο που τονίζει και τόνισε στην παρέμβασή του τη δυσκολία, την πολιτιστική και πολιτική που έχει ο πληθυσμός. Αυτή η ένταξη δεν μπορεί να γίνει αναγκαστικά με τη βία, με εμβριουλκό. Θα πρέπει ε, να το δέχεται ο πληθυσμός που από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας λέτε εσείς δεν ισχύει. Τα κριτήρια οικονομικής σύγκλησης πληρούνται. Είναι σαφές αυτό και αυτό οφείλεται στις πολύ σημαντικές προσπάθειες που έκανε η χώρα τα τελευταία χρόνια αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί. Προσοχή, προσοχή. Φυσικά, η Λετωνία σήμερα δεν είναι, σαν την Κύπρος. Θα ήταν πολύ απλουστευτική, πολύ απλοϊκή αυτή η σύγκριση. Αλλά πρέπει να προσέξουμε αυτό το κυπριακό σύνδρομο. Να μην κλείσουμε τα μάτια, να μην στρουθοκαμιλήσουμε. Γιατί δεν θέλουμε ο λύκος να μπει και να φάει τα πρόβατα θα πρέπει στην Ευρωζώνη τα κριτήρια να μην αποδυναμώνονται ούτω ώστε να δημιουργούνται νέοι φορολογική παράδεισοι. Τα ουσιαστικά υπόθηκαν από τους συναδέλφους μου και δεν έχουν προσθέσω πολλά για τις ρογμές που υπάρχουν, για τους κινδύνους που υπάρχουν, για τους οποίους θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Όλοι σας τονίσατε το θέμα της ρύθμισης του τραπεζικού μυστικού, του τραπεζικού απορρίτου, μπορεί η Λετωνία ε, εξ αυτού να γίνει ε, καταθετήριο ξένου βρώμικου χρήματος. Όπως είπατε και εσείς ε, κύριε Σεγητά, τα, οι μισές καταθέσεις είναι από ξένους. Κυρίως από τον μεγάλο γείτονά τους σε αυτή τη δεύτερη ρογμή. Θέλω να την υπογραμμίσω. Το φαντάζεστε κι εσείς. Υπάρχει και το θέμα της ε, φορολογικής στρατηγικής της κυβέρνησης της Λετωνίας που προσπαθεί να μειώσει όσο μπορεί τον εταιρικό φόρο και έτσι δημιουργεί σημαντική φορολογική στρέβλωση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Και έτσι θα, γίνει η Λετωνία ένα μικρό πλητήριο βρώμικου χρήματος. Και θα απορροφήσει ε, διάφορες εταιρείες που θα πάνε εκεί για λόγους α, φορολογικούς. Προσοχή λοιπόν, το ξέρετε πολύ καλά, το ψηφισμά σας, το ψηφισμά μας θα πρέπει να είναι το πολιτικό μήνυμα αυτής της επαγρύπνησης. Από τη συμφωνία μας, από τον ενθουσιασμό μας δεν θα πρέπει να παρεκκλίνουμε, αλλά θα πρέπει να επαγρυπτούμε παράλληλα και θα προτείνουμε ακριβώς κάποιες τροπολογίες ε, στο ψήφισμα, ούτω ώστε να ενισχύσουμε και άλλα συμπληρωματικά κριτήρια, ειδικά τα φορολογικά κριτήρια. Σας ευχαριστώ. Very indeed. On behalf... Και εμείς από την ECR. thank you, chairman, Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μεταφραστώ και να μιλήσω έτσι την ε, μητρική μου γλώσσα, τα λετωνικά. Θέλω, καταρχήν, να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω για, την, ε, για τον ενθουσιασμό, για τη θετική ατμόσφαιρα που έτσι πλαισιώνει τη Λετωνία κατά την ένταξή της στην Ευρωζώνη. Η πρόοδος μας είναι προφανής. Ε, η έκθεση σύγκληση της ΕΚΤ είναι καταφανής και σημειώνει την πρόοδο που έκανε η Λετωνία και οι διαφορές ως προς τη σύγκληση όλο και μειώνονται. Καταλαβαίνω βεβαίω τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι συνάδελφοι, ιδίως για την άποψη της κοινωνίας, της λετωνικής κοινωνίας. Μην νομίζετε ότι η κοινωνία δεν έχει, ο κόσμος, ο πληθυσμός δεν έχει αρκετές πληροφορίες. Ίσως ε, όλα αυτά τα αρνητικά νέα που κυκλοφορούν γύρω από το ευρώ καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν τον κόσμο και γι' αυτό υπάρχουν κάποιες ανησυχίες. Αλλά τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης υπερασπίζονται περισσότερο ή λιγότερο το ευρώ, αλλά κανένας δεν λέει ότι πρέπει να καθυστερήσει η ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη. Το τελευταίο εξάμεινο νομίζω ότι και η στάση του κόσμου βελτιώθηκε. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι το ευρώ θα σταθεροποιήσει και το χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας μας. Αλλά η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί. Και εδώ μιλάω για τις ξένες καταθέσεις κυρίως αλλά η υπηρεσία κεφαλαγοράς έχει αυξήσει τις προϋποθέσεις για τις κεφαλιακές απαιτήσεις και ποιοτικά και ποσοτικά και ένας από τους λόγους ε, για αυτή την αυστηρότητα ας πούμε είναι ότι η Λετωνία θέλει να ενταχθεί στο ευρώ. Αν λοιπόν μπλοκάρει κάποιος την πορεία της Λετωνίας προς το ευρώ νομίζω ότι αυτό θα είναι όχι προς το συμφέρον της ε, Ευρώπης. Η Λετωνία θα παραμείνει τόσο ή ευρωπαϊκή χώρα. Ε, με την ένταξή της, ε, οι διάφοροι κρατικοί φορείς θα συνεχίσουν απαρέγκλιτα τις προσπάθειές τους, γιατί είναι πολύ σημαντικό βεβαίως οι επενδύσεις των ξένων και των τρίτων χωρών ε, στη Λετωνία να πλησιώνονται, όπως υπόθηκε. Αυτή η δουλειά πρέπει να κάνουμε εμείς. Επίση, άλλο θέμα, ο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν συνεχίσουμε να ενισχύσουμε το χρηματοπιστωτικό τομέα και μόνο, δεν θα είναι καλό αυτό για τη Λετωνία. Εμείς καταλαβαίνουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε. Για την ενέργεια, για το χρηματοπιστωτικό τομέα, για τις τράπεζες και θα συνεχίσουμε τη δουλειά αυτή. Και τέλος. Με μεγάλη χαρά άκουσα την αξιολόγηση που μας κάνατε και ζητάω από τους συναδέλφους να υποστηρίξουν αυτή την, ε, ε, αυτό το κείμενο, αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστούμε κύριε Σίλε. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω και εγώ το γεγονός ότι υπάρχει λετονική διερμηνία στη σημερινή μας συζήτηση Υπογραμμίζω όμως ότι δεν υπάρχει ελληνική μετάφραση στην έκθεση του συναδέλφου. Αυτή είναι μια παρατήρηση διαδικαστική. Διότι επί της ουσίας και από το διάβασμα της έκθεσης και από την παρουσίαση του συναδέλφου η εκτίμησή μου είναι ότι κάνει ειλικρινή δουλειά, τίμια. Αυτά είναι τα δεδομένα, δεν οξοραίζει τις καταστάσεις και νομίζω ότι αποτυπώνει πραγματικά και επομένως είναι μια τίμια έκθεση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και στα αγγλικά που τη διάβασα και στα ελληνικά, αν υπήρχε μετάφραση, αυτή θα ήταν η εκτίμηση. Από εκεί και πέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να είμαι ειλικρινή. Ο, ο συνάδελφος το έβαλε κατά έμεσο τρόπο, ο συνάδελφο Κλίνς το έβαλε ευθέω. Πού να χαιρετήσουμε, ω τι να το χαιρετήσουμε το θέμα αυτό τη εισόδου τη Λετωνία στο ευρώ. ω μια νίκη του λαού ο οποίο δεν έχει ρωτηθεί, εν πάση περιπτώσει δεν έχει αποφανθεί, ή ως ένα απαραίτητο σημείο που χρειάζεται η ω ενα απαραιτητο διότι κλονίζεται, διότι έχει προβλήματα για να μην το πω δραματικά, διότι έχει την ανάγκη να φαίνεται ακόμα ελκυστική. Ή επιμέρους λοιπόν παρατηρήσεις, διότι πολιτικών παρατηρήσεων πρόκειται και το διατάφτα προς τα πού να πάει. Να πεις όχι τιμωρώ το λετωνικό λαό, δεν πρόκειται περί αυτού του θέματος. Ορισμένες λοιπόν παρατηρήσεις για πού συνθέτουν αυτό το, το, τη σκέψη. Πρώτον, σωστά λέει ο συνάδελφος, αυτά είναι τα κριτήρια του μάστρη. τα καλύπτει και με το παραπάνω η Λετωνία, τι παραπάνω θα έλεγε κανείς. Θέλεις αφού αυτά έτρεψαν τα κριτήρια. Ελάτε όμως που εδώ και είναι γενικότερο πρόβλημα όταν ευημερούν τα κριτήρια του Μάστριχτ, όταν πάνε καλά δεν σημαίνει ότι πάει καλά και η πραγματική οικονομία και η κατάσταση των ανθρώπων. Έδωσε στοιχεία ο συνάδελφο. Η Λετωνία, τρίτη φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 40% στο όριο τη φτώχεια. 15% ανεργία. 32% ανεργία των νέων. Δημογραφική μείωση. Μετανάστευση. Και άλλα που θα μπορούσε να πει κανεί, όχι ω μορφή στον λετωνικό λαό, ω αποτελέσματα μιας πολιτικής λιτότητας για το ξεπέρασμα της κρίσης. Επομένως η υπερκάλυψη των κριτηρίων, σωστά τίθενται αυτά είναι, δεν μπορεί να βάλουμε άλλα, σωστά τα αναφέρει ο συνάδελφος, έχει γίνει με το κόστος. Δεύτερη παρατήρηση. Εντάξει, μπαίνει η Λετωνία. Και αν ισχύει αυτό που είπαν άλλοι συνάδελφοι και ως ένα βαθμό το διοθέτω και εγώ. Εν τέλει είναι και μια πολιτική απόφαση εν τέλει είναι και μια πολιτική απόφαση για του λόγους δεν τους εστερνίζουμε, αλλά πάση περιπτώσει αυτή είναι η λόγη. Σήμερα με την εικόνα ή την εμπειρία που μας έδωσε η διαδικασία του ευρώ ότι εκεί όταν βρεθεί σε κρίση ο καθένας είναι μόνος του και η κάθε χώρα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση βλέπε Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρο τίποτα δεν αποκλείει αύριο η Λετωνία να μπει σε ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα λόγω των απαιτήσεων πρώτο, διότι θα ανακαλύψουμε ότι ο τραπεζικός του τομέας δεν λέω μια σειρά πράγματα που είναι γνωστά τι θα γίνει, τι γράφεται, τι δεν, είναι υπερδιογκωμένος. Ενδεχομένως να αρχίσουμε να ψάχνουμε ότι δεν δουλεύουν πολύ. Να πούμε ότι είναι και σπάταλοι και να μπει σε ένα καινούριο πρόγραμμα και τότε θα πούν δεν είναι σωστό να μπαίνει στην, Ευρωπαϊκή, στο στην Ευρωζώνη με πολιτικά κριτήρια, αλλά με οικονομικά. Κλείσαμε τα μάτια, το πληρώνουμε τώρα. Αχάριστοι αυτοί που του βάζουμε με αυτή την έννοια. Και αυτό έχει υποθεί σε πολλέ χώρε. Αυτό θέλω να επισημάνω και ο συνάδελφο, ξαναλέω, επί τη ουσία λέει τα πράγματα, δεν λέω εγώ τίποτα διαφορετικά στοιχεία. Και τελευταίο, για να μην σα ε, κουράζω, ο λετονικός λαός δεν έχει αποφανθεί. Δεν αμφιβάλλω ότι Εφόσον δεν υπάρχει ολοκληρωμένη ενημέρωση, δεν, δεν έχει πλήρη ενημέρωση. Το πρόβλημα όμως είναι εδώ. Γιατί αυτό το κριτήριο, κύριο Ρεν, το τι λέει η κοινή γνώμη σε σχετικέ ερωτήσει, το αποδοκίμασε. Λέει δεν μα ενδιαφέρει η κοινή γνώμη. Δεν είναι από τα κριτήρια του Μάστερ. Πράγματι δεν είναι. Δεύτερο, υπάρχει έτσι κι αλλιώ στην οικοδόμηση και τη Ευρωζώνη η αριστοκρατική αντίληψη. Κάποιοι ξέρουν το καλό ενό λαού, το βάζουν μέσα στην Ευρωζώνη κτλ. χωρί να το ρωτούν. Αλλά εντάξει, λέω είναι δημοκρατικό έλλειμμα, θα γίνει ενημέρωση, πιθανόν να, να γίνει έτσι πληθωριστική ενημέρωση υπέρ του ευρώ και να πιστούν οι Λετώνοι και κανένας δεν μπορεί να πει τίποτα. Αλλά όσο υπάρχει αυτό το έλλειμμα αγαπητοί συνάδελφοι και έχω εμπειρία από κάποια χώρα, δεν μπορείς μετά να ζητάς από ένα λαό που δεν ρωτήθηκε να πληρώσει συνέπειες για πολιτικές που δεν ρωτήθηκε αν είναι μέσα σε ένα πλαίσιο που εν πάση περιπτώσει τον ωφελούσε ή όχι. Εύχομαι να μην το συναντήσουμε στο μέλλον. Αν σα λέω διάφορε ζωφερέ καταστάσει, δεν εύχομαι αυτό. Τέτοιο μέλλον σε κανένα λαό, ούτε και στο λετωνικό λαό. Αλλά αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα το εξ αρχή, μετά το βρίσκει μπροστά ω ένα πρόβλημα και καμιά φορά δεν το βρίσκει με μορφέ που δεν θα ήθελε να το βρει. Και όχι με μορφέ συντεταγμένε, τούτο τ' άλλο κτλ. Αυτή λοιπόν η αισιόδοξη εκδοχή οικοδόμηση του ευρώ με αριστοκρατική όμως αντίληψη, δεν ρωτάμε, προχωράμε γιατί έτσι πρέπει να γίνει, εύχομαι να μην δημιουργήσει προβλήματα που βλέπουμε μπροστά μας στο λετωνικό λαό. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε κύριε Χουντή. Όπως είπαμε στα μέλη, υπάρχει ένα ειδικό γλωσσικό καθεστώς για αυτή την έκθεση γιατί ήταν πολύ περιορισμένη η ημερομηνία, η προθεσμία που είχαμε για την έγκριση. Έχουμε καταγγείλει ε, αυτή την απαράδεκτη ανεπάρκεια και την περιορισμένη προθεσμία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λυπούμε και εγώ για τις δυσκολίες που δημιουργεί. Τελειώσαμε με τους κοιόδης εισηγητές, περνάμε στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. and Mr. Ε, Mr. you have the floor. Uh, thank you very much. Uh, στα γερμανικά ο κύριος Κάρινς. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Μπάλτς για την καλή του έκθεση, για όσο και ισόρροπη. Μόνο 13 παραγράφους έχει. Νομίζω ότι πολύ εύκολα και γρήγορα μπορέσαμε όλοι να τη διαβάσουμε και τα όσα μας είπε εδώ ε, διήβριναν λίγο το πεδίο και μας ε, διαφώτισε και δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω όλα όσα είπε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάλτς. Και συνεχίζω στα αγγλικά λίγο τώρα. Uh, Ήθελα να σας πω, να κάνω κάποιες σκέψεις για το που είμαστε, όχι μόνο στη Λετωνία, αλλά και γενικότερα στην Ένωση, για τώρα και για το μέλλον. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική για την ε, συνοχή, την οικονομική συνοχή στην Ευρώπη. Στις βαλτικές χώρες υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση πέρα από την οικονομική. Για τη Λετωνία ε, αναφέρθηκαν διάφοροι ομιλητέ στην οικονομική διάσταση με μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια προς το νόμισμα θα τονωθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, οι επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ε, για τη Λετωνία και για άλλες χώρες ότι δεν έχουμε όλοι το ίδιο βιωτικό επίπεδο. Τότε που όμως πρέπει να αναρωτηθείτε, μα πώς διάολε να έχουμε όλοι υψηλό ε, βιωτικό επίπεδο αν δεν έχουμε τις κατάλληλες οικονομικές συνθήκες. Ε, το να είναι κανείς μέλος Ευρωζώνης είναι μια σημαντική διάσταση αυτού του εγχειρήματο. Επίσης να θυμίσουμε ότι η Λετωνία τα τελευταία πέντε χρόνια τελούσε, 50, 90 χρόνια τελούσε υπό ε, σοβιετική κατοχή και ε, δεν πρέπει να λησμονούμε την ιστορία και μετά από όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα το τελευταίο βήμα ε, είναι η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ και στην Ένωση τώρα θα μπει στην Ευρωζώνη και έτσι επιβεβαιώνεται ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας στον κόσμο το να είναι στην Ευρωζώνη μια χώρα δεν αρκεί ούτε για τη Λετωνία ούτε και για τις άλλες χώρες. Άμα ήταν το μαγικό ραβδάκι θα ήμασταν όλοι πολύ πλούσιοι, θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι και δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Δεν αληθεύει κανένα από αυτά τα επιμέρους στοιχεία, άρα δεν αληθεύει και το σύνολο. Αυτό που θέλουμε με την, Ευρωπαϊκή, με την Ευρωζώνη είναι να έχουμε ελεύθερη αγορά. Πρέπει να τονίσουμε και να ξανατονίσουμε την ε, σημασία της ενιαίας αγοράς. Ξέρουμε ότι κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών δεν είναι απολύτως ανοιχτή και αν έχουμε ε, την νομισματική ένωση χωρίς όμως να λειτουργεί πλήρως μία ε, ανοιχτή ενιαία αγορά δεν μπορούμε να αποκομίσουμε πλήρω τα ωφέλη ε, σε καμία χώρα. Δεν αξιοποιούμε το δυναμικό που υπάρχει. Και ποιο είναι αυτό το δυναμικό. Εμπορικές διαπραγματεύσεις ε, που αρχίζουν τώρα ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κομμάτι αυτού του δυναμικού, αλλά είναι ανόητο να ονειρευόμαστε τις ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές με τη ΣΥΠΑ αν δεν το έχουμε καταφέρει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε διάφορα εμπόδια στο δρόμο της επίτευξης της συμφωνίας ε, με την ΕΠΑ, αλλά πρώτα πρέπει να κανονίσουμε ε, να συμβεί αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, το πλέον σημαντικό ζήτημα είναι η νέα αγορά. Τώρα θα μιλήσω λετωνικά γιατί έχουμε και μετάφραση. Θα ήθελα να πω και κάποια πράγματα για αυτά που είπαν ε, οι συνάδελφοι για τον τραπεζικό τομέα και τις καταθέσεις ε, των ε, όσων δεν διαμένουν μόνιμα στη Λετωνία. Είπε ο εισηγητής ότι αυτό αντιστοιχεί στο 130% του ΑΕΠ. Είναι από τους μικρότερους τραπεζικούς τομέας. Ο μέσος όρος είναι 370% και οχταπλάσιο είναι, είναι ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου, Φερρυπίν. Ο μέσος όρος σας είπα είναι 370% και 800% στην Κύπρο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ε, τηρουμένο των αναλογιών είναι μικρός ο τραπεζικός τομέας και άρα δεν μπορεί να κλειδωνήσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όντως οι καταθέσεις κατά το 40% προέρχονται από μη κατοίκου τη Λετωνία. Αν ήταν ε, ε, ε, ε μεγαλύτερο ο τραπεζικό τομέα, αυτό θα ήταν ανησυχητικό. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, εποπτεύουμε την δραστηριότητα των τραπεζών που έχουν αυτές τις καταθέσεις, θεσπίζοντας υψηλότερες απαιτήσει ως προς τη ρευστότητα των τραπεζών και επίσης υπάρχει μια προθεσμία 30 ημερών αν δηλαδή αποσύρονταν όλες αυτές οι καταθέσεις πρέπει να κατοχυρώσουν οι τράπεζε ότι θα έχουν την ίδια ρευστότητα. Δεν είναι πολύ άριθμε αυτές οι τράπεζες. Ε, ε δεν χρηματοδοτούν την πραγματική λετονική οικονομία και είναι κάπως αποστασιοποιημένες από τον υπόλοιπο τραπεζικό τομέα που συναλλάσσονται με τις επιχειρήσεις. Τρίτον, για αυτές τις καταθέσεις ε, των όσων διαμένουν μόνιμα στη Λετωνία. Οι συναλλαγές γίνονται ως επιδοπλίστων σε αμερικανικά δολάρια και όχι ε, σε ευρώ. Οι τράπεζες λοιπόν αυτές που έχουν της εν λόγω καταθέσεις Οι ε, μάλλον όσοι έχουν καταθέσει σε αυτές τις τράπεζες έχουν αντίστοιχες καταθέσεις σε αμερικανικές τράπεζες. Σήμερα το πρωί συζητούσαμε το ζήτημα του ξεπλήματος, του βρώμικου χρήματος, της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων και το καθεξής. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ε, θα πρέπει να πλησιάσουμε κάπως ε, τις ε, αμερικανικές διατάξεις για αυτό το ζήτημα, διότι υπάρχουν πολλές αμερικανικές τράπεζες που συνεργάζονται με αυτές τις λετωνικές τράπεζες που έχουν τις εν λόγω καταθέσεις. Αυτές λοιπόν δεν συμμορφώνονται με τις αμερικανικές απαιτήσει. Έκλεισαν λοιπόν οι συνδεδεμένοι αμερικανικοί λογαριασμοί και υπήρχε εξοδικία. Δηλαδή ε, αυτές οι λετονικές τράπεζες έπρεπε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Αμερικανικού δικαίου διότι ήταν σε Αμερικανικά δολάρια οι συναλλαγές. Δηλαδή εποπτεύονται από τη Λετωνία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη ΣΥΠΑ αυτές οι τράπεζες. Ε, δεν είναι μια πάγια κατάσταση ε, και καταλαβαίνουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Σωστά είπε ο εισηγητής πως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταστήσουμε αυστηρότερες τις διατάξεις για την νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων. Αυτό είναι χρήσιμο για όλες τις χώρες και για όλες τις τράπεζες. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή. Thank you very much indeed, Mr. We give the floor. Σας ευχαριστούμε κύριε Κανίνς. Η κυρία Λούλινγκ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε ήθελα να πω στα γερμανικά στον κύριο Βάλτς ότι τον ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή του. Ε, το πολλό το F. Είναι πολύ καλή η έκθεση και συμπαγής. Ε, και τώρα στα γαλλικά... Θέλω να απαντήσω στον Έλληνα συνάδελφο, ο οποίος ε, παρενέβη. Ανησυχεί σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό της Λετωνίας. Για το κατά πόσον έδωσε τη γνώμη του. Εγώ θα, θα ήθελα να είχαν δώσει τη γνώμη τους και οι Έλληνες όταν εσείς ενταχθήκατε στο ευρώ, στην ευρωζώνη. Και θα ήθελα ο ελληνικός λαός να καταψηφίσει την ένταξη στην Ευρωζώνη, γιατί έτσι θα είχαμε πολύ λιγότερα προβλήματα όπως έχουμε τώρα. Εμείς Ε, δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Δεχτήκαμε κράτη-μέλη στο ευρώ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Η Ελλάδα είναι από αυτά. Υπάρχουν κι άλλα. Τώρα είμαστε πάρα πολύ επιμελείς, πολύ προσεκτικοί στο παρελθόν, της ε, στο παρελθόν με τη Λιθουανία ας πούμε, με διάφορα ερωτήματα. Θα ήταν, πολύ, θα ήταν πολύ πιο καλά εξοπλισμένη η Ευρωζώνη αν όλα τα κράτη που ανήκουν σε αυτή τώρα σεβόντουσαν τόσο καλά τα κριτήρια του Μάστριχτ, όπως το κάνει η Λετωνία. Μακάρι να ήταν σαν τη Λετωνία. η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωζώνης θα ήταν ευτυχής αν βρισκόταν στη θέση της Λετωνίας. Για να μην πω και η δική μου χώρα. Εγώ θυμάμαι τον ε, πρώην αδελφό σας, τον Ντομπρόφσκι. Και πρώην συναδελφό μα που ήταν εδώ. Ε, θαυμάζω αυτά που έκανε, αυτά που πέτυχε. Έκανε μεταρρυθμίσεις και όμω επανεξελέγει. Αν είχαμε κάποιον σαν γι' αυτόν σε όλε τι χώρε τη Ευρωζώνη, άτομα τα οποία δεν καταφέρουν να, κάνουν, να περάσουν τι μεταρρυθμίσει ή να τι περάσουν έγκαιρα, αν είχαμε τέτοια άτομα θα ήμασταν πολύ πιο ε, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις δυσχέρειες. Η κατάστασή μας είναι δυσχερής, Δεν μπορούμε να θέτουμε αυτά τα ερωτήματα για τη Λετωνία, δεν μπορούμε να, να τις δημιουργούμε δυσκολίες όταν τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δεν σέβονται αυτά τα κριτήρια. Για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τι λέγανε τα περισσότερα κράτη-μέλη, δεν θέλουμε να σεβαστούμε τα όσα μας λένε οι Βρυξέλλες, δεν, ξέρει τι λέει, δεν ξέρουν τι λένε αυτοί εκεί στις Βρυξέλλες κτλ. Αυτά είναι πολύ σοβαρά γιατί τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θέσπισαν όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και αυτό αφορά την ε, Ευρωζώνη. Όλα αυτές οι διαδικασίες αφορούν την Ευρωζώνη. Και ξαφνικά εδώ ξυπνήσαμε και έχουμε θέματα, ας πούμε, σε ό,τι αφορά την ε, ένταξη της Λετωνίας. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή από πού και ως πού. Επίσης, σε αυτούς που λένε ότι υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι λόγω των ξένων καταθέσεων. Ε, κοιτάξτε, Υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό. <laughs> Δεν είναι και καινούριο, έτσι. Ε, ε, λογικό είναι να υποφεληθεί η Λετωνία. Δεν απαγορεύεται. Είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, όπως και η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. το να βάζετε στο ίδιο καλάθι και να μιλάτε εδώ για τον κίνητο του να γίνει η Λετωνία φορολογικό παράδεισο είναι υπερβολικό. Σε ό,τι αφορά το τραπεζικό απόρριτο, η Λετωνία είναι μέλο τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα θέματα δεν αφορούν μόνο την Ευρωζώνη, αφορούν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Εγώ δεν έχω καμία ανησυχία. Σα το λέω. Αντίθετα. Και θα ήθελα να είναι κάποιο επικεφαλή Ευρωζώνη όπω ο κ. Ντομπρόφσκι που ξέρει από μεταρρυθμίσει ξέρει να τις επιβάλλει. Φυσικά ήταν δύσκολο για το λαό, αλλά το γεγονός ότι επανεξελέγει κάτι δείχνει. Είναι μια απόδειξη νομίζω ότι αυτός ο λαός είναι λογικός. Ότι ξέρει να διαφοροποιεί ανάμεσα στη δημαγωγία και σε αυτούς που πραγματικά υπηρετούν το λαό. Και πώς να το πω τώρα, ακόμα και αν υπάρχουν προβλήματα, ακόμη και αν πρέπει να καταπιεί κανείς το πικρό χάπι, το κάνει για τον καλό σκοπό. Είναι σε καλή κατάσταση σήμερα, είναι παραδειγματική, παραδειγματική χώρα και όλοι μπορούμε να διδαχτούμε. Νομίζω λοιπόν ότι περί των ανησυχούμε, καλό είναι να τους συγχαρούμε και να χαρούμε κι εμείς από αυτή την ένταξη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λούλιν. Και τώρα η κυρία Ντανούτα Χούμπνα. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ως Πολωνέζα, όταν μιλάω για τη Λετωνία φυσικά έτσι με σπρώχνει η ζήλια μου. Και θα ήθελα και η Λετωνία και η Ευρωζώνη να κερδίσουν από αυτήν την ιστορία. Αυτή η σχετικά χαμηλή υποστήριξη ε, χρήζει προσοχής, γιατί ξέρω ότι οι πολιτικοί ηγέτες στην Ευρώπη δουν ότι δεν υπάρχει υποστήριξη για την Ευρώπη, ας πούμε, δεν θα την ανέφεραν καν, γιατί φοβούνται, βέβαια, για την επανεκλογή τους. Γι' αυτό, λοιπόν, θαυμάζω το θάρρος της πολιτικής ηγεσίας της Λετωνίας. Όπως είπε και η κυρία Λούλινγκ, ο κύριος ε, ε, εξελέγει δύο φορές, επανεξελέγει δηλαδή. Όχι μόνο πρότεινε μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ε, είχε βάλει την Ευρώπη πολύ ψηλά στην ατζέντα του. Κέρδισε πολιτικά και τις εκλογές, αλλά από την άλλη υπάρχει αυτή η αντίφαση ότι υπάρχει χαμηλή υποστήριξη του ευρώ στη Λετωνία. Είναι πολύ σημαντική ενημέρωση. Γιατί νομίζω ότι η μικρή επίσημη υποστήριξη για την ένταξη στην Ευρωζώνη αντικατοπτρίζει την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης και το πώς θα μετατραπούν οι τιμές, οι μισθοί κτλ. σε ευρώ. Δηλαδή τα τεχνικά θέματα. Ε, Εκεί δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση και όλα αυτά θα πρέπει να εξηγηθούν επαρκώ στον ε, λαό. Τώρα, όπως είδαμε και από παλιές εντάξεις, ε, πολύ συχνά πρέπει να μπει κανεί στην Ευρωζώνη και μετά να αρχίσει να αυξάνεται η υποστήριξη για την ε, ανεργία. ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρώπη είναι 12,5%. Ε, είναι πιο ψηλό στη Λετωνία, αλλά όχι πάρα πολύ πιο ψηλό. Τέλο δεν είναι και ηλικιώδη, όπω η ανεργία σε κάποιε χώρε τη Ευρωζώνη. Ε, θα ήταν βεβαίω πολύ πιο ψηλή η ανεργία στην Λετωνία αν δεν υπήρχε μετανάστευση. Γιατί το γεγονό ότι υπάρχει μεγάλη μετανάστευση αποκρύπτει το πραγματικό πρόβλημα τη ανεργία. Όμω η ανεργία στη Λετωνία δεν ε, δείχνει μόνο το γεγονό ότι η κοινωνία αυτή ε, προσαρμόζεται και στην κρίση κτλ. Αλλά δείχνει και το βαθμό και το βάθος των ε, διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Θυμάμαι όταν η Εστονία εντάχθηκε. Μήνες πριν την ένταξη στην Ευρωζώνη, βλέπαμε την αντίδραση των αγορών. Τα σπρέντα έπεφταν και μειώνταν τα CDS. Ε, Όμω στην περίπτωση της Λετωνίας δεν βλέπουμε αυτή την εφορία των αγορών όπως το είχαμε δει στην ε, περίπτωση της Εστονίας. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Υπάρχει κάποιος λόγος γιατί δεν υπάρχει αυτή η θετική αντίδραση των χρηματαγορών για μια χώρα η οποία πρόκειται να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Σας ευχαριστούμε κυρία Χουμπνέρο, κύριος Γκίγκολ ε, ε, Σύντομος θα είμαι και εγώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάλτς για αυτή την έκθεση. Συμφωνώ με την ε, θετική προσέγγιση που έχει για την προσχώρηση στην Ευρωζώνη της Λετωνίας. Θα ήθελα και εγώ με σαφήνεια να πω προς τον συνάδελφο από την ΚΟΕ ότι οι Λετωνία έχουν κάνει την επιλογή τους για δύο λόγους και υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Όταν η Ελλάδα συζητούσε το ευρώ και πήραμε μια απόφαση, δεν υπήρχε το ευρώ πολύ καιρό ακόμη. Τώρα η Λετωνία μέσα από όλη αυτή την κρίση κρατήθηκε στο μηχανισμό, ε, δεν υποτίμησε το νόμισμα της, έκανε μάλιστα εσωτερική υποτίμηση για να μην απαγκιστρωθεί από το μηχανισμό ισοτιμιών. Και αυτό επιβαίνονται και πάλι με, την, με τις εκλογές. Οι Λετωνοί έχουν με δημοκρατικό τρόπο κάνει την επιλογή τους και όχι μόνο γι' αυτό αλλά επειδή χρησιμοποιούν το ευρώ σε πολλές υποαγορές είναι παρόν το ευρώ ήδη στη Λετωνία. Ρόμπερτ ε, μπορέσαμε ε, όταν επισκεφτήκαμε τη χώρα σου με την ΕΚΟΝ ε, να δούμε η δίσόμαση ότι υπάρχει ήδη το ευρώ. Λοιπόν, το θέμα πλέον έχει γίνει πολιτικό. Συμφωνώ με τον κύριο Κλίντς λοιπόν, και ο τρόπος ε, με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα στις βαλτικές χώρες και τώρα η Λετωνία η δεύτερη στη σειρά και είναι καταπληκτικό πώς κάνουν αυτή την επιλογή υπέρ της Ευρώπης και αυτές οι επιλογές είναι πολύ πιο ε, από, το, τότε, από την εποχή των τευτονικών υποτών. Ε, ε, είναι το αντίστροφο τώρα, μπαίνουν στην Ευρώπη και είναι πάρα πολύ καλό που κάνουν αυτήν την ε, συνειδητή επιλογή. Αλλά Παρότι είναι ξεκάθαρο όπως ε, βλέπουμε στην έκθεση του κυρίου Μπάλτς ότι πλήρει όλα τα κριτήρια η Λετωνία και το έχει αποδείξει με το μηχανισμό συλλαγματικών ισοτιμιών, ταυτόχρονα όμως υπάρχει ένα διανοητικό πρόβλημα. Θεσπίστηκαν τα κριτήρια τεκμέροντας βασικά ότι υπαρκούν αυτά τα βασικά ε, κριτήρια, ούτως ώστε να μην ε, καταρρεύσει η Ευρωζώνη. Δεν έχουν ε, τροποποιηθεί τα κριτήρια, όμως τώρα έχουμε διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, Έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα με τη δέσμη έξι οδηγιών. Και τώρα το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί δεν τροποποιούμε τα κριτήρια για την προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Φυσικά και εδώ θα συμφωνήσω και πάλι με την εκθέση του κ. Μπάλτς. Δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε ε, κάνει τα μαθήματά μας ε, και δεν έχουμε μελετήσει τα κριτήρια να τα αμφισβητήσουμε όλα. Το αντίστροφο πρέπει να κάνουμε και απευθύνω το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφόσον αλλάξαμε την νομοθεσία με τη δέσμη 6 οδηγιών, 2 οδηγιών και το νομοθέτημα για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες δεν επαρκεί αυτό ως λόγος για να αναθεωρήσουμε τα κριτήρια που θεσπίσαμε ακόμη και για την προσχώρηση νέων κρατών. Αυτό όμως δεν αλλάζει τίποτα στην αξιολόγηση για την Λετωνία. Πρέπει να αναρωτηθούμε εμείς αν είναι επικαιροποιημένα πλέον τα κριτήριά μας. Και η παρατήρηση πάλι σύντομη για τις ανησυχίες που υπάρχουν. Λοιπόν, έμαθα ότι είναι σχετικά μεγάλη η παραοικονομία στη Λετωνία και έχω κάποιους συνδυασμούς για αυτά τα συγκρίσιμα αριθμητικά στοιχεία. Πάλι σε εκείνη την επίσκεψη μάθαμε ότι ε, υπάρχουν θέσεις αποσχόλησης, αλλά όχι ε, καταγεγραμμένες. Ε, ως προς το μέγεθος τώρα του τραπεζικού τομέα. Πιστεύω ότι σε μια κοινή ενιαία αγορά δεν είναι ορθή πρακτική να πει κανείς ότι δεν μπορεί ε, τα ε, ξένα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο στο τραπεζικό τομέα μια ε, χώρα. Και συμφωνώ με αυτά που είπε η Άστριντ Λούλινγκ. Όταν έχετε ανοιχτή αγορά, δεν μπορείτε να αποφασίσετε ότι αυτές κάποιες χώρες δεν μπορούν να έχουν ξένα περιουσιακά στοιχεία πάνω από ένα ορισμένο ανώτατο όριο του ΑΕΠ τους όταν σε σχέση με την έκθεση Manival βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής των κανόνων περί νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων και αυτό ισχύει και για πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό πρέπει να μας ανησυχεί και πρέπει να μας ανησυχεί αν προετοιμάζουμε φορολογικά νομοθετήματα τα οποία... Ε, θα εποφελ... από τα οποία θα υποφεληθούν χώρες που θα μπουν στην Ευρωζώνη. Δεν συγκρίνω, δεν ταυτίζω τη Λετωνία με την Κύπρο, όμως αληθεύεται το 2011 ψηφίστηκε φορολογική μεταρρύθμιση στη Λετωνία, χάρη στην οποία εξαιρείται από τη φορολόγηση η διανομή μερισμάτων. Ε, αντίστοιχους κανόνες βλέπουμε σε φορολογικούς παραδείσους. Λοιπόν, ο φορολογικός συντελεστής ε, για τα εταιρικά κέρδη ε, είναι εξαιρετικά χαμηλός. Λοιπόν, όταν μιλάμε για μεγαλύτερη φορολογική ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το έχει ζητήσει επανειλημμένα, αυτό είναι προβληματικό, να έχουμε μια νέα χώρα η οποία ουσιαστικά τροποποιεί αντιστοίχως την φορολογική της νομοθεσία. Αυτό δεν ε, ε, σημαίνει ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε την προσχώρηση ε, της Λετωνίας. Όμως ε, ας αναρωτηθούμε, όλο ένα και περισσότερες χώρες υιοθετούν τέτοια φορολογική νομοθεσία για να είναι ελκυστικές από φορολογικής πλευράς και όχι επειδή είναι πραγματικά ανταγωνιστικές και με στοχευμένο τρόπο προσαρμόζουν την φορολογική της νομοθεσία για να προσελκύσουν αλλοδαπές επενδύσεις. Αυτή η διάσταση είναι πρέπει πρέπει να μας ανησυχεί και όπως είπε και ο συνάδελφος θα καταθέσουμε τις σχετικές τροπολογίες. Δεν πρέπει να χάσουμε όμως ένα θετικό πνεύμα που θα πρέπει να διέπει την ε, διαδικασία προσχώρησης της Λετωνίας στην Ευρωζώνη. Ευχαριστούμε Σβέν. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Χουντή και πάλι. Παρακαλώ όμως ε, να είστε λίγο σύντομος ε, διότι άλλα λίγα λεπτά έχουμε διερμηνία. the, the floor. Να είστε πολύ σύντομος. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και η κυρία Λούλινγκ να με ακούει τώρα. Αρκετοί συνάδελφοι απάντησαν ή μπήκαν στη συζήτηση που άνοιξε. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά γιατί η δημοκρατία έχουμε, ακούμε ο καθένα απόψει. Δύο-τρει παρατηρήσει όμω σε αυτά που είπε η κυρία Λούλινγκ Γιατί εκεί ήταν λίγο πιο αιχμηρά και ίσω και πιο προσωπικά. Πρώτο, λέει αποφασίσαμε ορισμένοι να βάλουμε κάποιου με πολιτικά κριτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη. Ερωτώ εγώ, ποιοι ποιοι αποφάσισαν να βάλουν κάποιους άλλους στην Ευρωζώνη με πολιτικά κριτήρια. Αλλά αν θέλετε το ερώτημα να πάει παραπέρα. Όσοι αποφάσισαν ή ισχυρότεροι να βάλουν ή να βάζουν κάποιους στην Ευρωζώνη το κάνουν ως φιλανθρωπική πράξη. Δείτε τα αποτελέσματα που αποκαλύφθηκαν με την κρίση. Στην Ευρωζώνη υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι πλέον και υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι ελληματικές. Συμπέρασμα, λειτουργεί κατά άδικο τρόπο. Δεύτερη παρατήρηση για να μην... Να ρωτηθούν όλοι οι λαοί. Ναι, να ρωτηθούν όλοι οι λαοί. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν το λέω ως υπεκφυγή. Να ρωτηθούν τη στιγμή που τίθεται το ερώτημα. Όχι τώρα που έγιναν κάτω από έναν εκβιασμό, λέει θέλετε εκλογέ, κάνετε κτλ. Και το τελευταίο, η τελευταία μου παρατήρηση. Προτρέπω, αν δεν έχει διαβαστεί, η έκθεση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα που λέει ότι με το πρόγραμμα και όλα αυτά ότι σώζεται η Ελλάδα, τελικά σώστε, εσώθη η Ευρωζώνη και όχι η Ελλάδα. Finish, τελείωσα, τελείωσα. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ please. που δώσατε το λόγο. Ναι, τελείωσα. τελείωσα. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, τελείωσα. Αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη λίγο να λέμε και καμία αλήθεια. Ή τουλάχιστον να λέω τη δική μου αλήθεια, όχι αυθαίρετα πράγματα όπως ισχυρίστηκε η κυρία Λούλινγκ ότι είπα. Ότι είπα αυθαίρετα. Thank very much indeed. Uh, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκίγκολτ ρώτησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να της δώσω ε, σύντομα το λόγο. Κύριε Λούλινγκ, σας παρακαλώ. Δεν είναι συζήτηση για την Ελλάδα, νομίζω. Ε, για τη Λετωνία συζητάμε τώρα. Ε, δύο λεπτά θέλω να δώσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει σύντομα στον κύριο Γκίγκολτ. Yes, uh, let me first... Ευχαριστώ. Θέλω να καλωσορίσω την ε, υποστήριξη για την ένταξη της ε, Λετωνίας στο ευρώ. Η Κομισιόν συμφωνεί με αυτά που ακούστηκαν στην, ε, στη συζήτηση και στην έκθεση ότι η Λετωνία πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες. προσπάθειες. Δεν τελειώνει εδώ η προσπάθεια, πρέπει να συνεχίσει με ισχυρές πολιτικές, συνετή δημοσιονομική πολιτική, ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγορά εργασίας κτλ. Είναι πολύ σημαντική η επίτευξη της Λετωνίας, αλλά δεν τέλειωσε εδώ η προσπάθεια. Από πλευράς Κομισιόν, να πω πολύ σύντομα ότι καταλαβαίνουμε πλήρως τις ανησυχίες που εκφράζει το Κοινοβούλιο για τη σύντομη χρονική περίοδο. Δεν γίνεται όμως πάντα κάτι καλύτερο. Ε, καταλαβαίνουμε και εκτιμούμε την ευέλικτη στάση του Κοινοβουλίου και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε στο μέλλον. Για τις παρατηρήσεις του κύριου Γκίγκολτ που αφορούσαν τους φόρους, όχι τα κριτήρια ένταξης και αν υπάρχει ανάγκη να τα αναθεωρήσουμε αυτά τα κριτήρια. Τα κριτήρια ένταξης αναφέρονται στη συνθήκη και φυσικά για να αλλάξουν πρέπει να αλλάξει η συνθήκη. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αν δείτε την αξιολόγηση της Λετωνίας, έχει το ποσοτικό και το ποιοτικό στοιχείο και διάσταση. Και η Κομισιόν και η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έκανε και τη δική της παράλληλη έκθεση, ασχολήθηκε πολύ με τη βιωσιμότητα της σύγκλησης. Δηλαδή όχι η σύγκληση μόνο τώρα, κατά πόσο είναι βιώσιμη αυτή η σύγκληση και δεν ε, βάλαμε σε κάποια κουτάκια απλώς. Βλέπουμε και το στόχο και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια συνολική εικόνα, μια σφαιρική εικόνα. Και όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα ε, με πείθουν ότι πραγματικά έχουμε μια σφαιρική εικόνα για την ένταξη της Λετωνίας. Είμαι θετικός, αλλά πάντα πρέπει να δίνουμε προσοχή και να κάνουμε μια υγιή, σωστή αξιολόγηση. Ο κύριος Κούτας και μετά ο εισηγητής μάλλον τώρα, ο κ. Μπάλτς. Πολύ σύντομα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όντως να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη χώρα και να παραμείνει σε αυτή τη συνετή γραμμή στην οικονομία της. Το έχω γράψει και στη δική μου έκθεση άλλωστε και χαίρομαι πάρα πολύ που γενικότερα το ενστενίζεστε. Ευχαριστώ για αυτό που είπε ο Βόλφ Κλίντς που στο μεταξύ αποχώρησε ότι το θέμα της ενέργειας θα πρέπει οπωσδήποτε να το έχουμε υπόψη μας και να το κοιτάξουμε. Τις τελευταίες εβδομάδες μου το έχουν αναφέρει πολύ Εγώ δεν μπήκα σε αυτό το θέμα γιατί ήθελα να κάνω μια μικρή έκθεση συμπαγή και συγκεκριμένη. Σε περίπτωση που θέλετε να συμπληρωθεί και να βάλουμε και την ενέργεια, με χαρά, είμαι πρόθυμος να το κάνω. Τώρα, τι θα... ήθελα να απαντήσω σύντομα. Είναι η ερώτηση, η προτροπή της Ντανούτα Χιούμπνερ. Γιατί μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται, δεν αντέδρασαν οι αγορές. Είναι γεγονός, με την Εστονία ήταν διαφορετική η κατάσταση ε, λίγο πριν μπει στο ευρώ, νομίζω οι αγορές περιμένουν να ληφθεί και επίσημα και τυπικά η απόφαση για ένταξη της Λετωνίας στην Ευρωζώνη και από εκεί και πέρα θα αντιδράσουν. Δεν έχω θορυβηθεί εγώ τώρα επειδή δεν αντέδρασε η αγορά. Ε, επίσημα δεν έχει ληφθεί απόφαση. Τους επόμενους μήνες θα το δούμε αυτό να σημαίνει. Ε, τελευταίο, αυτό που είπε ο Σπεν ακόμα και αν χρειάζονται τροποποίηση των συνθηκών, συμφωνώ απολύτως με την άποψή του ότι έχει σημασία να κοιτάμε και τα κριτήρια. Ισχύουν σήμερα με αυτή τη μορφή τα κριτήρια αυτά που είχαμε βάλει τότε. Γιατί. Υπάρχουν και τα κριτήρια του Γκέρτιγκεν και η νομική έτσι, απόφαση και κατάσταση, αλλά τα κριτήρια που είχαν θεσπιστεί τότε, ε, ε, μάλλον συγγνώμη, τα κριτήρια του Μαστρίχτ που ισχύουν τώρα, ε, ισχύ, ε, όπως ίσχυαν και στο παρελθόν έχουν την ίδια ισχύ. Σε αυτά τα κριτήρια βασίστηκα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Με χαρά να δω τις τροπολογίες σας και τις συμπληρώσεις σας σε περίπτωση που επιθυμείτε. Είμαι στη διάθεσή σας να τα εδώ όλα με επικοδομητικό και συνεργάσιμο ε, πνεύμα. Θα τα συζητήσουμε ξανά και την άλλη Δευτέρα είναι ψηφοφορία νομίζω. Ευχαριστώ κύριε ε, Μπάλτς, κύριε Γκίγκολτ σας είπα. Γιατί σας λέω Γκίγκολτ; πώς μου ήρθε. δεν πειράζει, δεν τρέχει γιατί. Μπάλτς. Καλά. Εντάξει, μέχρι Γκίγκολτ μπορείτε να με λέτε. Ε, λοιπόν, ε, χτες ε, ανακοινώθηκε ότι αύριο το απόγευμα στις, ε, αύριο στις 19 του μηνός λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες. Είναι πολύ επίγοντα όλα αυτά. 24 του μηνός θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα και θα ψηφίσουμε και ε, μάλιστα. Για να πάει τον Ιούλιο στην Ολομέλεια είναι κάτι επίγον το θέμα. Δεν έχουμε άλλα θέματα. Επόμενη συνεδρίασή μας τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι, 24 του μηνός στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση για την επόμενη συνεδρίαση.